Et la séance est reprise. Et la séance qui... Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι και ξεκινάμε, ξεκινάμε την ε, συνεδρίαση. L'appareil de vote électronique. Με ψηφοφορίες παρακαλώ. Βάλτε παρακαλώ την κάρτα σα ε, στο μηχάνημα για να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίζουμε δοκιμαστικά. Tout le monde a voté. Ψήφιστε παρακαλώ όλοι. Tout le monde n'a pas voté. Δεν ψηφίσετε παρακαλώ όλοι. Bon, eh bien, je vais considérer que vous avez tous voté. Θα θεωρήσω λοιπόν ότι ψήφισατε όλοι και θα κλείσω την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Avec une très forte majorité favorable. Πλειοψηφία υπέρ, λέει ο πρόεδρος. Avant d'aborder les questions à l'ordre πριν ξεκινήσουμε λοιπόν την ημερήσια κατάξη, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το εξής. Η συνεδρίασή μας εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμού έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και χρειαζόμαστε απαρτία λοιπόν, μιας και έχουμε ψηφοφορίες. Γιάν 4Q2 θα λάβει χώρα η συνεδρίαση εν λόγω. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αφού σας το υπενθύμισα λοιπόν και αυτό, να δώσω το λόγο στον κύριο Ντανιέλε Βιώτη, το Γενικό Εισηγητή μας, για το ψηφίσμα το οποίο και καλούμαστε να ψηφίσουμε όσον ούπο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να σας αναγγείλω κάποιες τεχνικές αλλαγές στο ψηφοφορία που είχε γίνει από τις 25-26 Σεπτεμβρίου. Μόνο μία ίσονο σημασία τεχνική διόρθωση που αφορά το κεφάλαιο 1α γαμή 04-03-05. Οι περισσότερες πληρωμές φτάνουν το 50% των νέων δεσμεύσεων, αλλά όσοι ξεπερνούν τα όρια του σχεδίου προπολογισμού θα είναι 873 67 ε, εκατομμύρια αντί για 884. Κατά τα άλλα, όλε οι γραμμέ που εγκρίναμε στο σχέδιο προπολογισμού για τι δεσμεύσει ε, θα χρησιμοποιηθούν και στι πληρωμέ. Αναλόγως θα προσαρμοστούν και τα κείμενα που θα ψηφιστούν τελικά. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Συγητά. Και τώρα περνάμε στις ψηφοφορίες. Έτοιμοι. Συμβαστική. Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συμβαστική 1 εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Οκτώ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική δύο. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Α, καταπίπτει. 16. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Συμβαστική, ε, συγγνώμη, τροπολογή 30 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά απόχες Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφοφορία ηλεκτρονική για την τροπολογία αριθμών 40. Εάν ψηφίσατε όλοι, πέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ισοψηφία. Απορρίπτεται ως εκ τούτου. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά. Πρώτο τμήμα, παρακαλώ. Πρώτο τμήμα 45. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Τη 45 καταπίπτει. 46 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 50 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58. Το ίδιο. 59 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 66 και 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Συγγνώμη. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ την 89. Περάς. Εγκρίνεται. 19 υπέρ, 14 κατά. 90 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 91 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 104, συγγνώμη. Ξεχωριστή ψηφοφορία για την 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Για την παράγραφο 49. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ την 108. Πέρας. Ισοψηφία 17 υπέρ, 17 κατά, απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος ζητείτε για την 115. Πέρας. Εγκρίνεται. Και ζητώ συγγνώμη. 116. Καταπίπτει, μιας και εγκρίθηκε 115. 117. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τον 117. Πέρας. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές ας κάνουμε παρακαλώ έλεγχο για την 127 πέρας Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά κιόλα. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άλλα τμήματα. 130. Υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά α, καταπίπτει 136 137 λοιπόν επίσης καταπίπτει ή όχι 138 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 145 υπέρ. Κατά. Υπέρ κατά. Ναι, αλλά να σηκώνετε τα χέρια σας λέει ο πρόεδρος. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν τον 145. Κυρία Γκάρντια Ζαμπάλ. Δεν ψηφίσατε. Ψηφίζουμε την 145. Μήπως υπάρχει κάποιο λάθος. Είμαι κατά της δικής μου της τροπολογίας. Πώς γίνεται. Πέρα της ψηφοφορία ε, ψηφοφορίας, λέει ο πρόεδρος, απορρίπτεται. 146, υπέρ. Κατά. Μερικοί σηκώνουν το χέρι, μερικοί όχι. Κουρασμένοι είσαστε. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 19-15 152 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 155 με την ε, προφορική τροπολογία του συγγετή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 24 προς 8. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα οι γνωμοδοτήσεις ε, των επιμέρους επιτροπών. Άφετ. Γνωμοδότηση Άφετ. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για την ΔΕΒΕ δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Στην Ήτρε, την 6 ψηφίζουμε. Ήτρε 6, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Κουλτ 9. Κουλτ 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 27 προς 5 και 2 εποχές. Συγχαρητήρια και η γενικά εισηγητά και σε όλους του Σκιώδης που συναντήθηκαν επανειλημμένως και χάρη σε αυτούς ετοιμάστηκε αυτός ο κατάλογος και οι συμβαστικές. Ευχαριστούμε και τη Γραμματεία και ευχαριστούμε και τον κύριο Ρούμπιχ. Διότι και εκείνο είναι συγητής για τα υπόλοιπα τμήματα. Ε, κακώς δεν σας ανέφερα και προηγουμένως. Και ανέφερα μόνο αυτού του γενικού εισηγητού. Και τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση Βάιντερε, σύσταση της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη. Ε, τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 και 19 μπορούν να ψηφιστούν μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 28 και τροπολογία 11 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 και 31 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ηλεκτρονική. Πέρας. Με μεγάλη διαφορά 27 προς 6 απορρίπτεται. 29 και 12 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση διότι δεν σηκώνουν όλοι τα χέρια τους άρχεται η ψηφοφορία 29-12 πέρας 7 26 ε, απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ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 Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αντιλογικές σκέψεις 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Για το σύνολο του κειμένου τροποποιήθηκε. Με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται 30 προς 3 και μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Βάιντερ. Τώρα έκθεση Howard. Θέσπιση του Διαστημικού πρόγραμματο τη Ένωση και του Οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Διαστημικό Πρόγραμμα. 2018. 18. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20. Υπέρ, 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εγώ τις κατάλαβα, αλλά να το απελευθεύσουμε. 20. Πέρας. Μπορούμε να ψηφίσουμε την τροπολογία Χολμαγέρ 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Α, δεν ψηφίσαμε την 6. Σωστά. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω, τέλος πάντων, να επαληθεύσουμε. 22. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε για το 12. Πέρας. Απορρίπτεται 24 προς 8. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά δεν είναι σαφές σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη 14. Πέρας. Εγκρίνεται. 18 προς 13. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. 16 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικός. 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 18 προς 12. 4 καταπίπτει. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται και για το σύνολο του κειμένου ως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. 30 προς 1 και 2 εποχές. Πρόταση Τόρβαλτς πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα μια σειρά από τροπολογίες, 37 έως 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5 και πρώτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μια σειρά από τροπολογίες 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23. Θα ψηφιστούν μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικός 42 πέρας Απορρίπτεται. 18 προς 14. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εταιρεολογικές σκέψεις 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να επεληθεύσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 20 προ 12. Ε, 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και στο σύνολο του κειμένου όμως τροποποιήθηκε. Α, δεν ψηφίσαμε την 4. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι, βλέπω γιατί. 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για το σύνολο του κειμένου, ω τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται αυτή. Εψήφισαν άπαντες. Πέρα. Έγκριση με 30 προς 2. Και το δεύτερο κείμενο του κυρίου Τόρβαλτ, Για την έρευνα και την καινοτομία. 5. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και έρχεται μια σειρά από το 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 και 2 που μπορούν να ψηφιστούν μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Α, κατέπεσε. Η 15 κατέπεσε. Παράρτημα. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για τις αντιλογικές σκέψεις. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρί... εγκρίνεται. 3 καταπεπτή, 4 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Για το σύνολο του κειμένου ως τροποποιηθήκε ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. Ψήφισαν άπαντε. Πέρας. Εγκρίνεται 30 προ 2. Συγχαρητήρια Νίλ Στόρβαλτ για τι δύο εκθέσει. σα. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση από την ε, Πορτογαλία για τη Λισαβόνα. Σε κάθε περίπτωση η Πορτογαλία είναι. Όλα μαζί. Για την έκθεση του Ζωζέ Μανουέλ. Ψηφίζουμε unblock. Όλες μαζί. Ένα. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και έξι. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για το σύνολο του κειμένου, ονομαστική ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. 29 προς 2. Συγχαρητήρια στο, Ζωζέ Μανουέλ. Θα δώσω το λόγο στον Γενικό Εισηγητή Σίκφριντ ε, Μούρεσαν για πέντε μεταφορές, πέντε εμβάσματα που προτείνεται να ψηφιστούν. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητή συνάδελφοι. Η πρώτη μεταφορά πίστοση είναι η απόφαση 21 τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, συνεπία τη έκθεση που έχει συντάξει ο συνάδελφο Φερνάντε, ε, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, 4,65 εκατομμύρια ευρώ για την Πορτογαλία. Νομίζω ότι ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντε έφτιαξε μια πάρα πολύ καλή έκθεση, την οποία προτείνω και να υπερψηφίσουμε λοιπόν 4,65 εκατομμύρια το αποθεματικό ε, στην κανονική ε, γραμμή για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι ο Γενικός Εισηγητής μπορεί να μας παρουσιάσει, λέει ο Πρόεδρος, και τις πέντε μεταφορές πιστώσεων. Δεύτερη απόφαση είναι η απόφαση 22 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Global Transfer, έτσι λέγεται, Κάθε χρόνο κάνουμε αυτή τη συνολική μεταφορά, λίγο πολύ σε αυτή τη χρονική περίοδο και μιλάμε για μεταφορά πληρωμών σε όλες τις κατηγορίες του προϋπολογισμού. Το συνολικό ποσό που προτείνεται φέτος είναι 952 εκατομμύρια ευρώ, 0,68% δηλαδή του ε, συνόλου των επιτρεπόμενων πληρωμών για τον προϋπολογισμό του 2018, 133 κονδύλια θέση του προϋπολογισμού αφορά αυτή η μεταφορά. Όπως και πέρυσι, ακριβώς τον ίδιο αριθμό έχουμε. Προτείνω κύριε Πρόεδρε να δοθεί ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει αυτή τη μεταφορά. Αν συμφωνείτε κι εσείς. Ναι, παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μουρεσάν ο Γενικό Εισηγητής σας ήδη σας ε, σκιαγράφησε την πρόταση για αυτή τη γενική μεταφορά Global Transfer 953 εκατομμύρια, λίγο περισσότερα το ποσό από το προηγούμενο. 680 ήταν πέρυσι, 850 ήταν πρόπερσι, αλλά γύρω πολύ ε, στα ίδια επίπεδα κινούμαστε. Θα ήθελα εν συντομία να κάνω ορισμένα σχόλια για τα πιο σημαντικά στοιχεία ανάγκα κατηγορία. Για το 1α προτείνουμε ενίσχυση συνολικά και οι βασικές γραμμές που θα ενισχυθούν είναι το Ταμείο Κίσων Εύση, 150 εκατομμύρια και τα δύο τελευταία χρόνια κάναμε το ίδιο. Προτείνουμε επίσης ενίσχυση του ΙΤΕΡ 148 εκατομμύρια μετά ε, την αναθεώρηση ε, τον Απρίλιο το 18 του baseline για το ΙΤΕΡ και επίσης ενίσχυση του Γκαλιλαίου που προτείνεται για ποσό 141 εκατομμυρίων. Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας, αυτού του τίτλου, έχουμε και κάποια ε, προγράμματα όπου έχουμε επιστροφή ε, κονδυλίων, όπως παραδείγματος χάρη σε κάποια κονδύλια για το Horizon 2020 και για την Ευρατόμ ε, και τα τρία σκέλη του Connecting Europe έχουμε κάποια ποσά. Τώρα για το 1Β Πολύ λίγα είναι τα κονδύλια εδώ. Ενίσχυση 3 εκατομμύρια για το πρόγραμμα υποστήριξη θρεπτικών μεταρρυθμίσεων. Πιο σημαντική είναι η κατηγορία 2, τίτλο 2, όπου εδώ προτείνουμε συνολικά ενίσχυση. Ενίσχυση συγκεκριμένα 150 εκατομμύρια για το πρόγραμμα αγροτική ανάπτυξη όπως απαιτείται με βάση τις ανανεωμένες εκτιμήσεις των κρατών μελών λόγω αυξημένη ε, ε, δυνατότητας απορρόφησης ε, σε ό,τι αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Κατηγορία τίτλος 3. Εδώ έχουμε κάποια προγράμματα που προτείνουμε να ενισχυθούν κυρίω το ΆΜΙΦ. 100 εκατομμύρια ευρώ και για 30 εκατομμύρια προτείνουμε να αυξηθεί το μέσο υποστήριξη την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις με την υιοθέτηση κάποιων νομικών βάσεων και γι' αυτό προτείνουμε επιστροφή χρημάτων για το σύστημα εισόδου-εξόδου και για το eu ΛΙΣΑ. Σε ό,τι αφορά τον τίτλο 4, εδώ συνολικά προτείνουμε επιστροφή κονδυλίων κυρίως από το ENI και το ΕΠΑ. E από το ENI προτείνουμε επιστροφή 187 εκατομμυρίων. Αυτό αφορά κυρίως καθυστερήσεις ε, στην εκπλήρωση των κριτηρίων για τη δημοσιονομική στήριξη και σε ό,τι αφορά ε, την... το ανατολικό σκέλος, η Μολδαβία και Ουκρανία και για τη νότια γειτονία Ιορδανία, Μαρόκο και Αίγυπτος. Τέλος, προενταξιακό πρόγραμμα, είπα. Προτείνουμε και εδώ 124 εκατομμύρια να επαναδιατεθούν, να, να κατανεμηθούν στο πλαίσιο αυτής της, παγκόσμια, της ε, γενικής μεταφοράς σε ό,τι αφορά τις γραμμές της Τουρκίας εδώ, τα κονδύλια που αφορούν την Τουρκία, δηλαδή που βλέπουμε ε, χαμηλούς ρυθμούς ε, ανάθεση συμβάσεων και εκτέλεσης ε, προγραμμάτων χαμηλότερες εκτιμήσεις από τα προβλεπόμενα μέχρι τα τέλη του έτους. Για να ολοκληρώσω, ε, κύριε Σιγητά, κύριε Πρόεδρε, και για να επαναλάβω αυτό το οποίο έχω προαναφέρει, σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα καταθέσει στην Επιτροπή σα πρόταση για μείωση των πιστώσεων πληρωμών όπω είχε γίνει το 2016 και το 2017. Επομένω, η υλοποίηση του προπολογισμού φαίνεται καλή και ελπίζω να μπορώ να βασιστώ στην υποστήριξή σας για τη γενική αυτή μεταφορά, το Global Transfer που θα μας επιτρέψει να έχουμε ε, εφαρμόσει, εκτελέσει πλήρως τον προπολογισμό μας μέχρι τα τέλη του έτους. Ευχαριστώ πολύ τον πρόσωπο της Κομισιόν, ο Πρόεδρος. Καλό είναι αυτό, γιατί αποφεύγουμε έτσι συσσόρευση υπολείπων προς εκαθάριση. Και ξέρουμε ότι είναι ένα πρόβλημα και οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί στο πλαίσιο του Πουδουπού. Έχετε εσεί ε, πληροφορίε να δώσετε, κύριε Μουρεσάνο, όχι δεν έχω ούτε ερωτήσει. Εγώ ε, θα πρώτα ψηφίσουμε υπέρ τη ε, γενική αυτή μεταφορά. Πάμε στι επόμενε. Τρίτη μεταφορά, απόφαση 23 τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προτείνει ενίσχυση, αύξηση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Διότι τα χρήματα αυτά χρειαζόμαστε για να πάει από το Λονδίνο στο Παρίσι ο οργανισμός λόγω του Brexit. 2,6 εκατομμύρια παραπάνω χρειάζονται και με βάση τους κανόνες για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το 60% προέρχεται από τις εθνικές εποπτικές αρχές και μόνο το 40% από εμάς, από το προπολογισμό της Ένωσης. Αυτό είναι ο για τον οποίο χρειαζόμαστε τα χρήματα από που θα τα πάρουμε, από πού θα τα πάρουμε από τον προπολογισμό που είχε διατεθεί για τον Ευρωπαϊκό ε, Οργανισμό Χημικών γιατί φέτος ε, έχουμε ε, μια, ένα πλεόνασμα 6 εκατομμυρίων ευρώ και επομένως μπορεί ε, να μεταφερθεί το ποσό. Άρα έχουμε συνολικά 1,6 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για να μετεγκατασταθεί από την έδρα της που είναι το Λονδίνο αυτή τη στιγμή στην έδρα στο Παρίσι και έπειτα έχουμε την απόφαση 24 του 2018 που αφορά ενίσχυση της εισφορά μας στην Ούντρα για το 2018 κατά, με το ποσό των 20 εκατομμυρίων σε πιστός ανάληψη υποχρέωσεων αλλαγή για τις πληρωμές δεν προβλέπεται. Γιατί χρειάζονται αυτά τα χρήματα, χρειάζονται διότι η Αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τη δική της εισφορά στην Ούντρα κατά 300 εκατομμύρια, όχι, συγγνώμη, 300 εκατομμύρια δολάρια. Και τώρα έχουμε ένα μεγάλο και μια μεγάλη τρύπα 270 εκατομμύρια δολάρια που χρειάζεται η ΟΝΤΑΡ για τις δραστηριότητές Από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα. Θα μειωθεί στη Γεωργία κατά 30 εκατομμύρια το ΕΠΑ. Έχουμε κάποια, εκεί, ε, κάποια κονδύλια από την Τουρκία, 2,8 από τις εισφορές που, που έχουν καταβληθεί στη στο Εθνικό Συμβούλιο Ζάχαρης, Ελιές ε, και τα λοιπά, 2,8 των Ευρωπαϊκών Πολιτικής Προστασίας 3 εκατομμύρια. Είχαμε προβλέψει μεγαλύτερο ποσό, μεγαλύτερες ανάγκες και 0,75 εκατομμύρια από τη γραμμή για την ετοιμότητα αντιμετώπιση ε, καταστροφών σε τρίτε χώρε. Το σχετικό ταμείο. Εκεί λοιπόν θα πάνε και από εκεί θα βγουν τα χρήματα. Ξέρω ότι υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται. Το έχουμε συζητήσει και προηγουμένως σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων που διδάσκονται τα παιδιά πρόσφυγες Παλαιστίνη. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα σχολικά εγχειρίδια θα εμπλωτιστούν με συμπληρωματικό υλικό και οι εκπαιδευτικοί ε, έχουν λάβει σαφείς οδηγίες να αντιμετωπίσουν τα θέματα, τα ζητήματα που προκύπτουν από μέρος περιεχομένου και έχουμε και την Ούνρα. Τα χρήματα που θα τις διατεθούν θα πάνε ε, στην ε, χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην πληρωμή των μισθών των ε, εκπαιδευτικών που διδάσκουν παιδιά Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Θα στηριχθεί λοιπόν η εκπαίδευση αυτή. Και πρέπει να σας πω ότι αν δεν διαθέσουμε αυτό το κονδύλι, οι δραστηριότητες της Σούντρα Επιτόπου θα κινδυνεύσουν θα σταματήσει εκπαίδευση, τα παιδιά αντί να είναι σε μια αίθουσα ε, διδασκαλία θα είναι στο δρόμο και καταλαβαίνετε τι κινδύνου συνεπάγεται όλο αυτό και για τη μετανάστευση και ενδεχομένω και για τη ριζοσπαστικοποίηση των παιδιών αυτών. Το θέμα λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω, των σχολικών εγχειριδίων το ε, συζητήσατε προηγουμένω σε μια συγκεντρία κυκλισμένων των ε, θυρών. Υπάρχει αποθεματικό για το του 2019, αλλά από αυτό το πλαίσιο και για τη μεταφορά ψώση το 2018, εγώ ψηφίσουμε κύριε Πρόεδρε υπέρ και τέλος έχουμε τρεις μεταφορές ε, με τις αποφάσεις 25, 26 και 27 αποφάσεις επιτροπής. Στόχος είναι μεταφορά 110 εκατομμυρίων σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 73 εκατομμύρια σε πληρωμές από το αποθεματικό των αναγκών και άλλες εκμεταλλευτήσεις ε, πιστώσει όπω πιλωτικά προγράμματα και προσπασκευτικέ ενέργειε. Πρώτον, για την Ιεμένη, απόφαση 25-5 εκατομμύρια ευρώ σε ανάληψη αποχρεώσεων και 32,5 σε πληρωμές για την ανθρωπιστική κρίση που έχει προκύψει και σοβεί στην χώρα. Για την αντιμετώπιση των βασικών πτυχών της κρίσης, τρόφιμα, υγεία, παροχή νερού, εκπαίδευση, ε, υγεία, τα βασικά, οι βασικές ανάγκες 50 λοιπόν σε ανάληψη υποχρεώσεων, 47,8 προέρχονται από το Emergency Aid Reserve και 2,2 από πιλωτικά προγράμματα και προσκευαστικές ενέργειες. Τέλο πάντων, ένα πιλωτικό προ και μία ε, προπαρασκευαστική ενέργεια που δεν μπορούν να εκτελεστούν. Οι μεταφορέ 31,3 από το Παναφρικανικό Πρόγραμμα λόγω κάποιων καθυστερήσεων 1,2 από το πιλωτικό πρόγραμμα και προσφαστική ενέργεια που ανέφερα πριν που δεν εκτελούνται Επομένως, προτείνω να ψηφίσουμε υπέρ της απόφασης 25 για την διάθεση του ποσού για την ΕΜΕ. Παρόμοια η 26 απόφαση για την περιοχή του Σαχέλ δεν δημιουργούνται προβλήματα. Το ίδιο ποσό 5 εκατομμύρια σαν λήψη αποχρεώσεων και 32,5 εκατομμύρια σε πληρωμές. Η απόφαση 27 αφορά τη λωρίδα της Γάζας 10 εκατομμύρια σαν αποχρεώσεων και 8 εκατομμύρια σε πληρωμές για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Λόγω της κλιμάκωσης ανθρωπραξιών και της βίας τους τελευταίους μήνες, τα χρήματα, ε, αυτά τα 10 εκατομμύρια σε ανάληψη υποχρεώσεων προέρχονται από το Παθηματικό Γενέκ της Ανάγκης και τα 8 από τη γεωγραφική συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ που έχουμε καθυστερημένη υλοποίηση κάποιων έργων και προγραμμάτων. Έχουμε λοιπόν χρήματα γιατί αναβλήθηκαν κάποια προγράμματα για του χρόνου. Αυτά τα τρία λοιπόν, ε, οι τρει τελευταίε πιστώσει, ε, μεταφορέ πιστώσεων δεν είναι καθόλου επίμεχε. Αυτά και ολοκληρώνω. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γενική Εισηγητά. Να ρωτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα μιλήσει για τα πολιτικά προγράμματα τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Είναι τα αγαπημένα των βουλευτών. Είναι ενθουσιώδης ε, όλοι. Τι γίνεται λοιπόν με τις πιστώσεις. yes, Chairman, uh, perhaps... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να διευκρινίσω να σας πω από τα 110 δισεκατομμύρια που προτείναμε για τις μεταφορές σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των πολιτικών προγραμμάτων και των προξενικών δράσεων μιλάμε για λίγο παραπάνω από 2 εκατομμύρια. Πρόκειται για ένα μικρό ποσό λοιπόν και πιστεύω ότι τα προπαρασκευαστικά, οι προπαρασκευαστικές δράσεις ε, για τις οποίες προτείνουμε τη μεταφορά έχουν παρουσιαστεί από τις ενδιάμενες εκθέσεις ως μη εκτελέσιμες. Άρα δεν προκαλεί, φαντάζομαι, αυτό έκπληξη στα μέλη της Επιτροπής σας. Πρόκειται ε, για τους νεαρούς Ευρωπαίους για την ανάπτυξη και το πρόγραμμα Υγεία για όλους. ένα πιλωτικό πρόγραμμα και μια προπροσκευαστική δράση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ερέλ. Ακούσατε το Γενικό Εισήγητη, κυρία συνάδελφοι. Ακούσατε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ευκρινήσεις της. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, κύριε Ντεπρέ. Μία ερώτηση ενημερωτικά, Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την μεταφορά, την μετακόμιση της αρχής τραπεζών. Βλέπω ότι το έξοδο θα τα επιβαρυνθούν 40% η Ευρωπαϊκή Ένωση και 60% η... τα κράτη-μέλη. Οι Βρετανοί δεν θα επιβαρυνθούν καθόλου, δεν έχουν μερίδιο. Θα δούμε και θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα και τα πορείσματα των διαπραγματεύσεων για το Brexit Έχουμε και την Επιτροπή Ελέγχου των Προπλαγισμών, έχουμε την κυρία Γκρέσλε μαζί μας, αλλά ως τώρα τα πράγματα έχουν μείνει στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως θα μπορούσε ο κύριος ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας διαφωτίσει. Κύριε Ντεπρέ. σε ό,τι αφορά το 40% για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 60% από τις εθνικές αρχές, αυτή η αντιστοιχία, αυτό το ποσοστό ισχύει και για τον ΕΟΠΑ και για το ΕΜΠΑ και για την ΕΣΜΑ. Πρόκειται λοιπόν ε, για ε, ένα ποσοστό το οποίο ισχύει εφάπαξ και τις τρεις ε, υπηρεσίες. Είναι ο κανονικός κανόνας δηλαδή που ισχύει για όλες τις υπηρεσίες αν το Ηνωμένο Βασίλειο α, συμφωνήσει, θα συμμετέχει κατά 60%. Στο 60% οι Βρετανικές αρχές θα συνεισφέρουν. Θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν ε, ε, στο 60% αυτό. Ναι, κύριε Ντεπρέ, αυτό που λέτε ότι το 60% είναι η συγχρηματοδότηση αλλά δεν αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βασίλειο αποφάσισε. Άρα, αν θα πρέπει να υπάρχει άλλο ποσοστό ενδεχομένω και το παράπλευρα αυτά, τις παράπλευρες αυτές απώλεια. Πρόεδρε, ο κ. Ζέλστρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε το λόγο. Μία ερώτηση έκανα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη νομική σχέση γιατί προβλέπει η συνθήκη ε, σε περίπτωση αποχώρηση ενό κράτου μέλους βασί του άρθρου 50 και αν υπάρχει ε, έντρα υπηρεσία στο κράτος αυτός. Ε, είναι επιτακτική ανάγκη μετακόμιση της υπηρεσίας και ποιο επιβαρύνεται με το κόστος. Ήταν σαφή η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πουθενά στη συνθήκη και στα πρωτόκολλα δεν προβλέπεται νομική υποχρέωση μετακόμισης της υπηρεσίας. Θα μπορούσε λοιπόν η υπηρεσία να βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η απάντηση που με έδωσε πριν από έξι μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση το Συμβούλιο είναι αυτό που αποφάσισε ότι χρειαζόταν, ήταν απαραίτητη η μετακόμιση. Άρα θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργη αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Κόλμελα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μπορεί να έχει περάσει και η ώρα και να έχουμε κουραστεί. Και τώρα προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από το Brexit με τη μετακόμιση μια υπηρεσία. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρουμε, γιατί πάρα πολλά θέματα είναι κρεμή και ανεπίλητα. Όσο και να επιμένουμε, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε στην παρούσα φάση. Ο προεδρό. νομίζω ότι καλά θα κάνουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή. Είναι τμήμα των διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η συνέχεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα να σας ε, καλέσω να αποφανθείτε επί τη μεταφοράς αυτής σε 21 με ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Μπορούμε να ψηφίσουμε και unblock όλες μαζί στις ε, ψηφοφορίες, στις ε, τροπολογίες. Για αυτές τις 7 μάλλον ε, μεταφορές, συγγνώμη. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. «22 υπέρ, δύο κατά, συγχαρητήρια» στον εισήγητη για τις υπόλοιπους, τα υπόλοιπα τμήματα και τις μεταφορές για τον προϋπολογισμό του 2018. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία τροποποίηση έχω να σας πω και πέντε μεταφορές. Καταρχάς, το συνέδριο που ζήτησε μετα... να μετατραπεί μία μόνιμη θέση σε προσωρινή θέση προκειμένου να διευκρινίσουμε ότι δεν χρειάζεται ψηφοφορία και εγώ υποστηρίζω το αίτημα αυτό, δεύτερο αίτημα σε ό,τι αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών που έκαναν αποταμίευση σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις και τις μεταφράσεις. Προτείνεται λοιπόν αυτό το αποθεματικό να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους. Καταρχάς, να καλέσουν περίπου 100 νέους πολιτικούς από την περιφερειακή διάσταση σε, στην 8η διάσκεψη πολεών και δήμων του χρόνου και κατά δεύτερον να καλέσουν το website, την ιστοσελίδα για τα κοινωνικά ε, μέσα εν ώψη και των ευρωεκλογών. Εγώ το υποστηρίζω και αυτό το τιμά λοιπόν. Τρίτο θέμα. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τέσσερις μεταφορές, δύο εκ των οποίων θα απαιτούσαν ψηφοφορία. Η πρώτη έχει να κάνει με τα μεγαλύτερα έξοδα συντήρησης και έχουν ε, γίνει διάφορες αποταμιεύσεις από διάφορες υποδομές τεχνικές 4,2 ε, εκατομμύρια ευρώ. Αυτό πρέπει να το ψηφίσουμε και συστήνω να ψηφίσει η Επιτροπή μας υπέρ. Δεύτερη, μικρότερη μεταφορά μετά από πρόορη σύνταξη προς το συμφέρον της υπηρεσίας υποστηρίζω και τα χρειάζεται ψηφοφορία. Τρίτη, μεγάλη μεταφορά για να αυξηθεί η χρηματοδότηση της ε, μετάφρασης γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Εδώ βρήκαμε πόρους σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις από το Πουδουπού και λόγω διαφορών καθυστερήσεων. 3 εκατομμύρια ευρώ είναι η μεταφορά. Αυτό θέλει πάλι να το ψηφίσουμε. Και εγώ πάλι είμαι υπέρ. Τελική μεταφορά. Προσωπικό ασφαλείας ε, συγκεκριμένα. Και χρειαζόμαστε 3 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για επιπλέον προσωπικό και πάλι μικρή μετατόπιση ε, προσωπικού. Δεν χρειάζεται εδώ ψηφοφορία στο κεφάλαιο αυτό, στο τμήμα αυτό και πάλι εγώ είμαι υπέρ. Άρα έχουμε δύο ψηφοφορίες για τη μετάφραση και για τη συντήρηση των κτηρίων. Ευχαριστώ κύριε Σίτα. Να στραφώ προς τους κοιότης. Έχετε να κάνετε ερωτήσεις, σχόλια. Όχι. Πολύ ωραία. Δεν ζητά κανείς το λόγο. Άρα η μεταφορά 5 και 6 θεωρούνται εγκεκριμένε εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Είστε σύμφωνος? Μάλιστα. Στο 5 και στο 7 μπορούμε να κάνουμε μία και μόνο ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, έναρξη. Tout Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. «23 υπέρ ψήφοι, δύο κατά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Κυρία Χόλμαϊερ, δεν ε, έχει οποιοδήποτε αίτημα σε ό,τι αφορά τα κτίρια. Και άρα, συνάδελφοι, νομίζω ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτή την μεγάλη και ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πολύ άρεθμοι από την αρχή μέχρι το τέλος και να σας υπενθυμίσω ότι στις 6 ε, και 4 έχουμε ραντεβού για την κοινή συνεδρίαση και μιας και κανείς άλλος ζητάει τον λόγο, πέρα στη συνεδρίαση.